Il Presidente. Care colleghe, cari colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ξεκινάει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την επιδημία ισχυρή και ακόλη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Επίτροπο Ντάλι για πέντε λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις σε σχέση με την επιδημία αυτή. Ανησυχώ για το υψηλό ποσοστό θανάτων και ασθενειών που προκάλεσε η επιδημία αυτή στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε αυτούς οι οποίοι υποφέρουν από αυτό. Θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται. Υπάρχουν άνω των 2.670 περιπτώσεων και υπάρχουν σοβαρές επιπλοπές, ε, επιπλοκές σε 660 περίπου ασθενείς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν προκληθεί 21 θάνατοι στη Γερμανία και ένα στη Σουηδία. Σποραδικές περιπτώσεις έχουμε και σε 11 άλλες χώρες και η Ελβετία έχει αναφέρει 15 περιπτώσεις και 4 έχουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες το επίκεντρο της ασθένειας είναι η περιοχή του Αμβούργου στη Βόρεια Γερμανία. Οι περισσότερες περιπτώσεις εκτός Γερμανίας αφορούν πάντα είτε Γερμανούς πολίτες οι οποίοι ταξιδεύουν, είτε πρόσωπα τα οποία έχουν επισκεφθεί αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της Γερμανίας. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την επιδημία αυτή. Πρώτον, αμέσως ενεργοποιήσαμε όλα τα δίκτυα που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση κρίσεων. Τα δίκτυα αυτά επικοινωνούν συνεχώς, ανταλλάσσουν πληροφορίες και ανοίγουν τον χώρο για να υπάρξει δυνατότητα ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε συναντήσεις με τις υπηρεσίες της αρμόδιες για την υγεία για να εξετάσει την εξέλιξη της επιδημίας τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και την θεραπεία των ασθενών. Το σύστημα ε, προειδοποίησης στον τομέα των τροφίμων είναι μια σταθερή βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών. Δεύτερον, ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών να προχωρήσει σε μια επιστημονική μελέτη η οποία ενημερώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της επιδημίας. Έχουμε τώρα έναν σωστό καθορισμό της περίπτωσης την οποία έχουμε μπροστά μας που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση πιο αποτελεσματικά. Ερωτηματολόγια συγκεντρώνονται συνεχώς και εξετάζονται από την ε, αρμόδια κοινοτική αρχή η οποία κάνει συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές στον τομέα της υγείας σε όλες τις χώρες και υπάρχουν φυσικά και στο, ε, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις υπηρεσίες των κρατών μελών και στις ε, επαγγελματικές κατηγορίες που ασχολούνται με την επιδημία αυτή. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε ε, μια διαδικασία η οποία μειώνει το χρόνο εξέτασης ενός δείγματος για να δούμε αν υπάρχει το εσκερίχια κόλλη από έξι ημέρες σε δύο ημέρες μόνο. Σε καθημερινή βάση έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές προστασίας των τροφίμων και ελέγχου των τροφίμων στις διάφορες χώρες. Θα ήθελα να ζητήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν ε, τις επιστημονικές μόνο ανακοινώσεις προς το κοινό έτσι ώστε να μειωθούν οι αδικαιολόγητοι φόβοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις διάφορες υπηρεσίες της συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τα Υπουργεία των διαφόρων χωρών για τον έλεγχο της επιδημίας. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται να προχωρήσουμε στον έλεγχο της πηγής της μόλυνσης. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η προσπάθεια. Ζήτησα από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της, του Συμβουλίου Υγείας χθε να ενισχύσει τον έλεγχο και τα μέτρα τα οποία παίρνει έτσι ώστε να εντοπιστεί η πηγή ε, της ασθένειας αυτής, της μεταδοτικής αυτής ασθένειας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λοιπόν άμεσα οι αιτίε αυτή τη μόλυνση. Οι γερμανικέ αρχέ δέχτηκαν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει στη Γερμανία εμπειρογνώμονε στον τομέα τη επιδημιολογία και ασθενειών που μεταφέρονται και προκαλούνται από τα τρόφιμα και από την ΕΦΣΑ. Στις, θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου οι εμπειρογνώμονες τις προσπάθειες αυτές για την επιδημία και θα συνεισφέρουν στις προσπάθειες ανείχνευσης της πηγής όπως γνωρίζουμε οι αρχικές υποψίες ότι υπεύθυνα ήταν τα αγκουράκια από την Ισπανία δεν επιβεβαιώθησαν από ιεσδήποτε δοκιμές και ελέγχους. Στις 15 Ιουνίου, στις 5 Ιουνίου ανακοίνωσαν οι γερμανικές αρχές ότι επί τη βάση των ελέγχων πιθανώς οι φύτρες σόγιας να είναι κάτι το οποίο προκάλεσε την πηγή που επηρέασε την κατάσταση άσχημα στο βόρειο τμήμα της Γερμανίας. That is also on my mind, but then uh, The information was Οι πληροφορίες αυτές απεστάλησαν άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις Ζώτροφες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις πάρα πολύ προσεπτικά και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες την στιγμή που έχουμε επιπλέον, ε, επιπλέον πληροφορίες. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοιες επιπλέον πληροφορίες θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές αρχές να μην βιαστούν, να δίδουν πληροφορίες για τις πηγές μόλυνσης οι οποίες δεν έχουν αποδειχθεί πλήρως από βακτηριολογικές αναλύσεις γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο διαδίδει αδικαιολόγητους φόβους στους πληθυσμούς της Ευρώπης και δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στους παραγωγούν τροφίμων οι οποίοι πολλούν τα προϊόντα τους στην Ένωση αλλά και εκτός Ένωσης. Εντατικέ έρευνες λοιπόν συνεχίζονται, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην καταλήγουμε σε πρόωρα συμπεράσματα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίε πληροφορίε από την Γερμανία σχετικά με την πιθανή πηγή ε, φύτρα. Τα τεστ δεν έχουν ολοκληρωθεί, οπότε ε, κάποια πρόωρα συμπεράσματα πρέπει να αποφευθούν. Αυτό δείχνει την σημασία που παίζουν τα κράτη-μέλη τα οποία όταν θα πρέπει να δίδουν στοιχεία στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης να είναι τα στοιχεία τους αυτά έγκυρα, τεκμηριωμένα, αποδεδειγμένα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα και προσοχή. Μπορούμε λοιπόν να μάθουμε από το τι συμβαίνει και να βελτιώσουμε τα συστήματά τους. Επαναλαμβάνω, το σύστημά μας λειτουργεί. Θα πρέπει να βγάλουμε τα κατάλληλα μαθήματα και συμπεράσματα. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων μας να είμαστε ευέλικτοι αλλά και ταχύς στα πλαίσια της ρύθμισης των διαδικασιών που ακολουθούμε για ανταπόκριση σε τέτοιου είδους συμβάντα. Ο συντονισμός και η σωστή πληροφόρηση και επικοινωνία είναι ο πυρήνας της ικανότητάς μας να είμαστε αποτελεσματικοί σε τέτοιες καταστάσεις. Θα πρέπει να πάρουμε ό,τι μαθήματα γίνεται στον τομέα αυτό. Δύο επιπλέον σημεία πριν κλείσω. Πρώτον, σχετικά με τις πιθανότητες απαγόρευσης και ορισμένων προϊόντων, κυκλοφορίας ορισμένων προϊόντων. Σας θυμίζω ότι το πρόβλημα ε, εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή γύρω από την πόλη του Αμβούργου. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα με τις προσπάθειες λοιπόν πιστεύουμε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων τροφίμων θα ήταν δυσανάλογη. Είμαι ευαίσθητο επίση και στις οικονομικές επιπτώσει που η κρίση είχε και έχει στους παραγωγούς οποροκυπευτικών κυρίω. Γι' αυτό συνεργάζομαι πάρα πολύ στενά με τον Επίτροπο Τσίολο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας οι οποίοι χτυπήθηκαν από την κατάσταση αυτή. Σήμερα γίνεται ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και μόλις τελειώσω θα επιστρέψω στις Βρυξέλλες για να συναντηθώ με τον συνάδελφο Τσίολος και θα είμαι παρόν σε αυτό το έκτακτο Συμβούλιο Γεωργίας. Ταυτόχρονα είμαστε σε συνεχή επαφή με τρίτες χώρες και με τη Ρωσία έτσι ώστε να τους πείσουμε να καταργήσουν την απαγόρευσή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες λοιπόν με ένα στόχο να τερματιστεί η επιδημία αυτή το ταχύτερο δυνατόν και επιμένω σε όλους τους εμπλεκομένους ότι σε τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε όχι με αντίληψη τοπική, εθνική αλλά ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και ευχαριστώ και για την πληρέστατη παρουσίαση που μας κάνατε. Ξεκινούμε με τους αγωγητές των πολιτικών ομάδων. Πρώτον, πρώτα δίνω το λόγο στον κύριο Πίτερ Λίζε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ντάλι, που καταρχήν έσυψε το βλέμμα του προς τους ασθενείς και θα ήθελα να το κάνω και εγώ το ίδιο. Εκατοντάδε ατόμων είναι βαριά άρρωστα. Το ιατρικό προσωπικό στη Βόρεια Γερμανία αμήνεται μέχρι τα όρια. 22 άτομα έχουν ήδη απαθάνει και χθε στο Συμβούλιο ο εκπρόσωπος ενό κράτου μέρους του Λουξεμβούργου είπε στο Συμβούλιο χθε ότι το οικονομικό, η οικονομική ζημιά διορθώνεται, η ανθρώπινη ζημιά όμως όχι. Και γι' αυτό ακόμα και αν δεν ξέρουμε 100% ποια είναι η πηγή, αν έχουμε κάποια υποψία, οι πληροφορίες αυτές ε, λέγεται πρέπει να γίνουν δημόσιες. Θα πρέπει να βρούμε όμως και την πραγματική ε, πηγή και με την υποστήριξη της ΕΣΑ γίνεται αυτή και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Τέλη που βοηθάν στην ε, ε, εξερεύνηση. Και εγώ όμως ως Γερμανός βουλευτής δεν μπορώ να πω όλα πάνε καλά. Υπήρξαν κάποια προβλήματα. Παραδείγματος χάρη η γερουσιαστής υγείας του Αμβούργου ενημέρωσε την κοινή γνώμη για τα ισπανικά αγγούρια δικαίως παρόλο που δεν ήμασταν σίγουροι Πρώτα ενημερώθηκε όμως η κοινή γνώμη και μετά αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ισπανικές Αρχές. Αυτό δεν ήταν σωστό. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας ότι ο εχθρός δεν είναι η Ισπανία ή η Γερμανία. Ο εχθρός είναι το βακτηρίδιο αυτό. Και στην ε, περασμένη σύνοδο της Ορομέλης εξετάσαμε το θέμα της αντίστασης ε, στην αντιβίωση. Εδώ έχουμε πραγματικά την ίδια περίπτωση ότι αυτός ότι εδώ έχουμε μία αντίσταση στα, ε, στην αντιβίωση και θα πρέπει να εργαστούμε στην την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο που σας δίδεται. Η κυρία Μακάβαν τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχετε δίκιο, Επίτροπε. Το θέμα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και θα έπρεπε τώρα να αντιμετωπίζουμε τους ασθεν... τα πρόβλημα των ασθενών και να εντοπίζουμε την πηγή. Αλλά πώ θα σταματήσουμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πριν από λίγε μέρε, συνάντησα κάποιους εκπροσώπους ε, τη ε, Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και μου, αναφερό... μου, ανέφεραν τα ζητήματα της ε, ασθένεια αυτής στι ΗΠΑ όταν αυτό δεν είχε εμφανιστεί στην Ένωση. Τώρα με την επιδημία θα έπρεπε να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Μήπως είναι οι αγροτικές πρακτικές που ανέφερε ο κ. Λίζε, είναι η εντατική καλλιέργεια των κυπευτικών είναι η χρήση, η υπερβολική χρήση αντιβίωσης στα ε, ζώα ή την ε, διασπορά κοπριάς. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ταχύτερα την πηγή της μόλυνσης. Ξέρω ότι λείπει το Συμβούλιο εδώ, αλλά το Συμβούλιο αρνείται να βάζει επισήμανση χώρας προέλευσης στα τρόφιμα. Μέχρι τώρα ελπίζω αυτό να αλλάξει στις συζητήσεις στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα κύριε Επίτροπε και να ενσωματώσουμε στις πολιτικές μας την πρόληψη. Προσφέρουμε πολλοί από εδώ στο σώμα ε, αναδιαφέρονται μάλλον πολλά για την υπερβολική νομοθέτηση αλλά συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις βάζουμε μπροστά τις ανάγκες τη αγοράς και όχι τις ανάγκες της προστασίας της υγείας και του κανολωτή. Προφανώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με business as usual και απλά να μην τρώμε σαλάτες. Χρειάζεται να αλλάξει πολιτική στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μακάβεν. Η κυρία Κορίν Λεπάζο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που μιλήσατε για τα θύματα και τους ασθενείς πρώτα. Πραγματικά αυτούς πρέπει πρώτα να σκεφτούμε μαζί με τους γεωργούς που είναι επίσης μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες που καταλαβαίνουμε απόλυτα. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, υποστηρίζουμε την αρχή της προφύλαξης. Εφαρμόστηκε ε, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να παραπονεθούμε. Πρέπει βεβαίως να αναλάβουμε και τις συνέπειες. Προτεραιότητα, το υπενθύμισε ο κύριος Λίζε, είναι οι άνθρωποι. Πριν το οικονομικό ζήτημα που μπορούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώ ο θάνατο είναι οριστικό. Δεύτερον, συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Μακάβαν. Πόσο σπουδαία είναι η ανιχνευσιμότητα. Σήμερα συζητούμε την επισήμανση. Είναι θεμελιώδε να είναι πλήρη η επισήμανση με πλήρη ανιχνευσιμότητα για να ξέρουμε από πού προέρχεται το προϊόν. Τρίτον, το εξαιρετικά ουσιαστικό θέμα της πηγής του προβλήματος. Ας δεχθούμε ότι δεν ξέρουμε τα πάντα, ότι υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, να δεχθούμε ότι μερικές φορές αγνοούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να αμφισβητούμε όσους παίρνουν αποφάσεις και να λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε. Εδώ πρέπει να υπερισχύσει η αρχή της προφύλαξης. Ευχαριστώ κύριε Λεπάζ. Ο κύριος Νίκολσον για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω ότι συμπάθειά μου προς όσους επλήγησαν και τα συλληπιτήρια σε όσους έχασαν τη ζωή, στις συγγενείς, συγγενείς έχασαν τη ζωή τους. Πιστεύω ότι δείχνει η κατάσταση ότι δεν είναι σωστό να καταλήγουμε σε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Καταλαβαίνουμε την οργή της ισπανικής πλευράς και όσων έχασαν ε, οικονομικά, αλλά η ζωή είναι αυτό που μετράει, γιατί τη ζωή δεν μπορεί να τη φερει πίσω. Έχουμε μία στέρεη βάση απάντησης, το είπε και ο Επίτροπος. Πρέπει να υπάρξει επίλυση της παρούσης κατάστασης το συντομότερο δυνατό και μακροπρόθεσμα να βελτιώσουμε την δυνατότητα ανταπόκρισής μας σε παρόμοιες περιπτώσεις. Εύκολα μπορεί να πει κανεί τώρα τι θα έπρεπε να είχε γίνει, τι δεν θα έπρεπε να είχε γίνει. γνωρίζοντα τώρα την κατάσταση. Θα πρέπει ωστόσο να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και σωστά το είπε ο επίτροπο, Πρέπει να δράξουμε μαθήματα από τη σημερινή κατάσταση. Πάντα μαθαίνει κανείς από τα λάθη του και αυτό θα πρέπει να γίνει και τώρα. Ευχαριστώ. Για δυόμιση λεπτά η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σωστά είπατε ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλοί νεκροί και ασθενείς από τα βακτήρια αυτά. Θεωρώ ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε καταδεικνύει ότι ούτε η Γερμανία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένες για μία ε, εξάπλωση του βακτηρίου ε, η σύγκριση με άλλες χώρες ε, καταδεικνύει ότι θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι. Θα σας δώσω εδώ το παράδειγμα των ΙΠΑ που από τη δεκαετία του 80 και εδώ υπάρχουν τεράστιες προσπάθειες στην έρευνα υποχρέωση δήλωση, συγκέντρωση των αρχών καταπολέμησης στην Ατλάντα που έχει πάρα πολλές ε, δυνατότητες και παρέμβασης όταν ξεκινήσει μια τέτοια επιδημία. Στη Γερμανία των Αντώνων έχουμε δύο ε, υπουργεία που είναι υπεύθυνα και δεν μπορούσαν καν να συμφωνήσουν ποιος, είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Έχουμε επίσης τα ομοσπονδιακά κρατήδια που πρέπει να αναλάβουν ευθύνες ε, και που τους ξεπερνάνε οι απαιτήσει αυτές Έχουμε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των εργαστηρίων και των πολιτών, πολιτικών, συγγνώμη, πότε δηλαδή θα πρέπει να δράσει η πολιτική και πότε θα πρέπει να παρέμβουν τα επιστημονικά εργαστήρια. Καταλαβαίνω ότι αν ε, σε μία υπουργό φτάνει το μήνυμα ότι φταίνουν τα αγκούρια θα προειδοποιήσει κατά αυτόν. Αλλά πού είναι η πραγματική αρμοδιότητα για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη μου δίνεται εντύπωση ότι με τις φύτρες, και το λέω πολύ προσεκτικά, και με τις φύτρες υπήρχε πολυφορική βία σύνη, όπως και με τα αγκούρια. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε να είναι υποχρεώση δήλωσης κεντρικά στην Ευρώπη, να υπάρχουν κεντρικά εργαστήρια και κεντρική υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε περίπτωση μιας τέτοιας επιδημίας. Μια υπηρεσία που θα έχει και την ε, αρμοδιότητα και εξουσία απόφασης. Ευχαριστώ τον κύριο Λίζε που αναφέρθηκε στα προβλήματα της αντιβίωσης και αυτό είναι κάτι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ότι πρόκειται για ένα γνωστό πρόβλημα. Επειδή όμως εμείς φοβούμαστε την συζήτηση με τον ιατρικό ε, τομέα, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τη μαζική εκτροφή Γι' αυτό δεν κάνουμε καμία συνεπή συζήτηση για την αντίσταση στα αντιβιώτικα. Γιατί έχουμε εδώ ένα πραγματικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαμπίν Βίλς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η επιδημία αυτή καταδεικνύει τα συστηματικά συστήματα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην απελευθερωμένη εσωτερική αγορά τροφίμων τη Ευρώπη. Αν το κέρδος προηγείται της προστασία των ατόμων, αυτό βλέπετε τι σημαίνει. Λόγω του βακτηρίδιου του ΕΤΕΚ πέθαναν στην ε, Γερμανία μέχρι στιγμή 22 άτομα και υπάρχουν πάνω από 1500 ασθενεί. 600 ασθενείς είναι ασθενούν πάρα πολύ ε, βαριά και έχουν ε, και το κίνδυνο νευρολογικών συνεπειών. <clears throat> Δύο εβδομάδες μετά που ξεκίνησε το αποτέλεσμα είναι ακόμα ασφαλής <clears throat> γιατί αν είχαμε μόνο τοπική εξάπλωση των τροφίμων θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ανοιχνευτεί η πηγή. Λόγω όμως της ε, μεγάλων αποστάσεων μεταφοράς τους και των ανωνύμων προϋποθέσεων παραγωγής δεν μπορεί να τηρηθεί η ανιχνευσιμότητα. Η ανιχνευσιμότητα όμως είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ξέρουν πού παράγονται τα τρόφιμα που τρώνε και πώς. Η Ομοσπαϊκή Κυβέρνηση Γερμανίας απέτυχε παντελώς στην αυτή την περίπτωση. Λόγω της ε, διαφωνίας αρμοδιοτήτων μεταξύ ως κρατηδίων και κεντρικής κυβέρνησης δεν μπόρεσε να γίνει τίποτε. Δεν ήταν προετοιμασμένη για μια τέτοια περίπτωση. Χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση της αγιορικής πολιτικής. Θα πρέπει τα τρόφιμα να είναι ασφαλή. Θα πρέπει όμως και οι παραγωγοί να προστατευτούν από ε, ε, προβλήματα απρόβλεπτα σαν αυτά εδώ. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν καθαρή και απαραίτητη αποκέντρωση της παραγωγής των τροφίμων και της διάδοσης αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σώσα Βάγνερ, 1,5 λεπτό. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, Τρει παρατηρήσει για την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε σχέση με τα ε, αγκουράκια. Είμαι γονό Γερμανού, αγαπώ τη χώρα. Είναι προφανέ, ωστόσο ότι οι γερμανικέ αρχέ αντέδρασαν βεβιασμένα και χωρίς φρονιμάδα. Επίσης, αν εξετάσουμε την ευρωπαϊκή αντίδραση διαπιστώνουμε ότι η ασφάλι, η επιτροπή και οι υπεύθυνοι αντέδρασαν με ασαφή και ε, καθυστερημένο τρόπο. Δεν μπορούσαν ούτε να συντονίσουν ούτε να, να κατευθύνουν. Τρίτον, οι, όσοι ζημιώθηκαν πρέπει να αποζημιωθούν γρήγορα. Αυτή τη στιγμή προτείνω το κοινοβούλιο, στο Κοινοβούλιο να οργανώσουμε στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο εδώ μια μεγάλη επίδειξη ευρωπαϊκής γαστρονομίας που θα βασίζεται ακριβώς στο ο Χάινριχ Μπέλ έλεγε ότι πρέπει να αποκτήσουμε, να ανακτήσουμε τη χαμένη τιμή. Η Ευρώπη είναι ο χώρος για να ανακτήσουμε τη χαμένη τιμή των Ισπανών Γεωργών. Ευχαριστώ κύριε Σώσα. Η κυρία Εράντς Γκαρσία, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτον, είναι υποχρεωτικό να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας για τους 23 νεκρούς στη Γερμανία και τη Σουηδία. Η κρίση δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ το σύστημα εσωτερικού συντονισμού για τα θέματα τροφίμων. Τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη έδειξαν βραδύτητα, αναποτελεσματικότητα και Ακόμα, μετά από 23 νεκρούς, δεν μπορούμε να πούμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα προβλήματα που, δημιουργούν, που δημιουργούνται από την αδράνεια σε παρόμοιες περιπτώσεις ή από τη βεβαιασμένη αντίδραση σε άλλες και την οικονομική, τις οικονομικές συνέπειες καταστροφής θέσεων ενεργασίας, ανεργίας και υγειονομικής κρίσης βέβαια με σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού. Ενώ στην Επιτροπή ε, εκφράζατε ή απειχούσατε τις ανεύθυνες εκφράσεις ε, γερμανικών ε, υπευθύνων δίνοντας ονόματα και επώνυμα ε, Ισπανών γεωργών ο γερμανικός πληθυσμός υφίστατο τις συνέπειες του βακτηρίου και ενώ νόμιζαν ότι ήταν ασφαλείς έτρωγαν κάτι που μπορεί να τους έβλαπτε η Επιτροπή θα πρέπει σήμερα να πει στο Συμβούλιο Γεωργίας την εξής πρόταση να χρησιμοποιηθούν τμήμα από τα 2,5 δις που υπάρχουν ως υπόλοιπα, μην χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα της, ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής, τμήμα αυτό να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και να βρουν ένα νομικό τρόπο να γίνει κάτι τέτοιο. Το βρήκαμε και σε άλλες περιπτώσεις και για τις διοξίνες και για την ΣΕΒ. Κύριοι Επίτροποι, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Υπουργοί, σήμερα στο Λουξεμβούργο πρέπει να σταθείτε στο ύψος των ευθυνών σας. Επιπλέον, οι γερμανικές αρχές μετά τις ε, ανεύθυνες δηλώσεις τους θα πρέπει εξ αρχής και αδιαμφισβήτητα να υποστηρίξουν αυτή, αυτό το μέτρο και να χρηματοδοτήσουν με δικά τους κονδύλια εκστρατείες ε, ενημέρωσης και ε, ευαισθητοποίησης υπέρ των προϊόντων που ε, υπέστησαν αυτές τις ζημίες. Ο κύριος Καπούλας Σάντους για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η επιδημία η οποία ξεκίνησε στη Γερμανία μας ε, οδήγησε θα έλεγα σε μια δύσκολη περίπτωση διαχείρισης κρίσης. και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαχειρίστηκαν τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε να κάνουμε με μια ανθρώπινη τραγωδία με δεκάδε νεκρού, με κινδύνου για τη ζωή εκατοντάδων άλλων και που θέτει στην επιφάνεια, φέρνει στην επιφάνεια ε, τα προβλήματα στην κυκλοφορία των προϊόντων των τροφίμων. Η κοινότητα θα πρέπει να δώσει μια ταχυτάτη απάντηση για τις αιτίες της κρίσης και τότε μόνο θα υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση της. Βέβαια οι συνέπειες προκαλούν και παράπλευρες απώλειες και αναφέρομαι στους παραγωγούς οποροκυπευτικών. Ήδη μίλησαν συνάδελφοι για αυτούς και πράγματι κατηγορήθηκαν εντελώς αδικαιολόγητα και τα εισοδήματά τους έχουν πλέον καταστραφεί. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε έτσι ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις στο μέλλον να μην επαναληφθούν. Καλό θα ήταν να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας της χρήσης αντιβιωτικών στα ζώα, σαν παράδειγμα. Ένας άλλος τομέας θα μπορούσε να είναι η νέα μορφή οργάνωση της ΚΑΠ. Και η βοήθεια που θα δίδεται στο μέλλον θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την αηφορία και την ποιότητα των παραγωμένων προϊόντων. Ευχαριστώ κύριε Κάπουλα Σάντος. Ρίς ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 23 είναι τα θύματα και άνω των 2.000 ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εντοπίσουν πράγματι με αποτελεσματικό τρόπο την πηγή της επιδημίας. Από την άλλη λοιπόν τα λαχανικά ο κόσμος τα περιφρονεί τώρα πλέον και δημιουργήθηκαν προβλήματα όχι μόνο υγιεινής και υγείας αλλά και κοινωνικά οι παραγωγοί οποροκυπευτικών αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και θα συνεδριάσουν γι' αυτό και οι Υπουργοί Γεωργίας στο Λουξεμβούργο σήμερα το απόγευμα. Πέρα από ό,τι ακούσαμε για την ανιχνευσιμότητα και την αρχή της πρόληψης, το θέμα είναι πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία που οδήγησε στην καταδίκη των Ισπανικών αγκουριών χωρίς καμία απόδειξη θα πρέπει το σύστημά μας ε, να βασίζεται ε, σε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες επιστημονικές ε, ανακαλύψεις και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννος Βοησισόφσκι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την αλληλεγγύη μου προς τις οικογένειες των θυμάτων. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ ταχυτά ανάρρωση σε αυτούς οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από την επιδημία. Δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε τις πηγές της επιδημίας αυτής μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε επίσης ε, καταφέρει να αντιμετωπίσουμε και τις πηγές των στρεβλών πληροφοριών που κυκλοφόρησαν σε όλη την Ευρώπη. Δημιουργήθηκαν τεράστιες οικονομικές ζημίες και παρανοήσεις ακριβώς εξ αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι αιτίες πρώτα που προκάλεσαν την επιδημία αυτή. Κυρίως θα πρέπει να δούμε ε, ποιες είναι οι χρήσεις αντιβιωτικών ε, στις μεγάλες κτηνοκροφικές εγκαταστάσεις. Γιατί αν χρησιμοποιούν τα αντιβιωτικά πράγματι σε τέτοια μαζική κλίμακα, τότε δεν θα πρέπει να μας εκπλήσουν τέτοιου είδους φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα πρέπει να περιορίσουμε λοιπόν στο μέγιστο την χρήση των αντιβιωτικών στην εκτροφή των ζώων. Χάουσλινγκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η επιδημία αυτή δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι όπως και στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προετοιμασμένη απέναντι σε μια τέτοια κρίση. Τρεις εβδομάδες χρειάζονται μερικές φορές για να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί και αυτό είναι απαράδεκτο. Τα οικονομικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να έχουν την πρωτοκαθεδρία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιος κηρύσσει ε, την κατάσταση, θα έλεγα, έκτακτης ανάγκης και ποιος τη διαχειρίζεται από εκεί και πέρα. Στη Γερμανία τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Υπάρχουν δύο, δύο ομοσπονδιακά υπουργεία τα οποία είναι υπεύθυνα, δημιουργούνται προβλήματα γι' αυτό και οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να εμπλακούν πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω τελικά αν βγάλαμε τα απαιτούμενα συμπεράσματα από τις κρίσεις στα τρόφιμα στη δεκαετία του 90. Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, απαιτείται εφαρμογή της αρχής της ανιχνευσιμότητας, απαιτείται μια σωστή επισήμανση των προϊόντων και απαιτούνται επίσης δυνατότητες παρέμβασης ιατρικά ασωστές. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Φεραίρα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενώπιον αυτή τη μεγάλη σειρά νέων για το θέμα αυτό, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάποιε πρακτικέ παρατηρήσει. Πρώτον, 15 μέρε μετά την εμφάνιση της ασθένειας και ένα μήνα μετά την πρώτη εμφάνιση κρούσματος, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση δεν λειτουργεί σωστά. Δεύτερον, είναι σοβαρή περίπτωση, αλλά δεν είναι απομονωμένη. Μην ξεχνάτε την πρόσφατη συζήτηση που είχαμε για τις διοξίνες. Οι περιπτώσεις είναι δείγματα μιας κοινή γεωργικής πολιτικής που έχει στόχο να προωθήσει την εντατική εξαγωγική καλλιέργεια και όχι την προστασία του καταναλωτή με καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα. Επίσης, οι γεωργοί της Ευρώπης όχι μόνο στο Νότο που πλήττονται, αλλά παντού πρέπει να προστατευθούν και να υπάρξουν μέτρα ούτω ώστε η κοινή γεωργική πολιτική να καλύψει τις ανισότητες που υπάρχουν. Ο κύριος Νίκ Γκρίφιν τώρα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Πρώτα ήταν τα αγκούρια. Χθε ήταν οι φύτρες. Τώρα δεν είναι οι φύτρες. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρουν τίποτα. Γίνονται κατα... κατηγορίες που καταστρέφουν οικονομίες και ζωές. Ξέρουμε όμως κάτι πολύ παράξενο. Ότι υπάρχει ένας ε, ένα μια παράξενη δομή του DNA στον, ε, στο βακτήριο αυτό. Επί, ε, σε πολλ... είναι ισχυρότερο από, μια, από ένα σύνηθε κρούσμα και δεν μπορεί να βρεθεί σε ένα ή δύο, σε μία ή δύο σειρές αλυσίδας τροφίμων. Σε πολλές χώρες, Βρετανία, Ιράκ, Ισραήλ, Ηνωμένε Πολιτείε, αναφέρθηκαν ότι χρησιμοποιείται ως βιολογικό όπλο μια γενετικά των τροφιμων ή κολλή. Μήπως αυτό είναι ένα, μια δοκιμή δοκιμή σε ζωντανή πραγματικότητα ενός βιολογικού όπλου. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Η επιδημία αυτή παραμένει μυστηριώδης. Προφανώς εκφράζουμε τη θλίψη μας για τους νεκρούς. Αυτό απαιτεί ωστόσο αυστηρότητα στην αντιμετώπιση ζητημάτων δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και χρειάζεται να συνεργαστούμε με ερευνητέ και φαρμακευτικές εταιρείες για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε μια τέτοια κατάσταση. Το βακτήριο στοιχίζει ζωές, πολλές ζωές, στοιχίζει και πολλά χρήματα στους γεωργούς και υπονομεύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στη γεωργική παραγωγή και την ε, γεωργοδιατροφική βιομηχανία που είναι η πιο ελεγχόμενη ωστόσο και ασφαλέστερη στον κόσμο μετά τα αγκούρια, τις τομάτες, τις, τις, τα μαρούλια και τις σόγια. Ποιος θα υπολογίσει τα ψυχιο, τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης λειτουργήσε πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ωστόσο ότι η Κομισιόν δεν έχει ούτε τα μέσα ούτε τη δυνατότητα να ελέγξει την αληθοφάνεια των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη-μέλη. Σήμερα τα βακτηρίδια κυκλοφορούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Άρα χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία και καλύτερη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης. Απαιτείται να υπάρχουν ε, καλύτερη χρησιμοποίηση των εμπειριών και, και επιπλέον ε, έλεγχοι πριν δεχθούμε οποιαδήποτε συμπεράσματα μιας ε, εθνικής ή περιφερειακής υγειονομικής αρχής. Επιπλέον, η κρίση δικαιολογεί απόλυτα την ενίσχυση της ανιχνευσιμότητας των τροφίμων, την υποχρέωση αναφοράς τη χώρα ένδειξη ή του τόπου προέλευσης στα τρόφιμα, κάτι που δεν προβλέπεται σήμερα παρά σε περιορισμένες περιπτώσεις δυστυχώ. Θα έπρεπε να επεκταθεί η υποχρέωση αυτή σε ένα μεγαλύτερο αριθμό τροφίμων που θα επέτρεπε να εντοπίζουμε ταχύτερα και κλείνω σε περίπτωση ε, κρίσης διατροφής την πηγή προέλευσης και να προλάβουμε την επιδείνωση της κατάστασης. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ. Ο κύριος Γιώλα Άινεν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι γεωργοί μπορεί να αποζημιωθούν. Δεν μπορούμε όμως να αναστήσουμε τα θύματα. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήρια προς τις οικογένειες όλων των ε, ατόμων που έχασαν τη ζωή τους και, τα και την ευχή ανάρρωσης όσοι είναι ασθενείς. Τρεις εβδομάδες μετά το ξεκίνημα της κρίσης δεν γνωρίζουμε τα αίτια. Πιστεύω ότι στην Ένωση είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν να μάθουμε πολλά πράγματα από αυτό, από αυτή την κατάσταση. Πρώτον, πού είναι η πηγή της επιδημίας. Είναι απαράδεκτες πρακτικές στην παραγωγή τροφίμων ή στην, αλυσίδα, στην διατροφική αλυσίδα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ένωση μια νομοθεσία που έχει ηλικία 20 ετών και ένα δίκτυο με εξαιρετικά υψηλά στάνταρ ασφάλειας. Πλην όμως βλέπουμε ότι η Ένωση είναι ακόμα ευάλωτη. Για τα τρόφιμα υπάρχουν προφανώς κενά ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν. Επίσης συμφωνώ με όσους είπαν ότι το θέμα της επικοινωνίας ήταν χαοτικό. Η επικοινωνία δεν πέρασε. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη Ευρώπη, το είπαν πολλοί συνάδελφοι. Ε, αν, το αν κάθε φορά μια περιφερειακή υγειονομική αρχή ξεκινήσει συναγερμούς, μπορεί να οδηγηθούμε σε περίπλοκες καταστάσεις, όπως συνέβη. Διαπιστώνω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο σύγχρονο και καλύτερο σύστημα με υποχρέωση κοινοποίηση και καλύτερης ενημέρωσης της κοινή γνώμης. Η κυρία Παρβάνοβα, ένα λεπτό. Η Γερμανία και οι ευρωπαϊκές αρχές προσπαθούν να βρουν ποιες είναι οι πηγές αυτής της μόλυνσης, αλλά δεν έχουμε ακόμα αρκετές αποδείξεις. Όλα τα σενάρια λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ακόμα και η πιθανή σκόπιμη χρήση και εισαγωγή του βακτηρίου αυτού στην τροφιμική αλυσίδα. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω τις ανακοινώσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις ανακοινώσεις ε, των γερμανικών αρχών όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες. Δεν είναι η πρώτη φορά ε, που έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και γι' αυτό θα πρέπει οι γερμανικές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην ανιχνευσιμότητα των προϊόντων. Η διαφάνεια απαιτείται έτσι ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στα τρόφιμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα κυκλοφορούν οι πληροφορίες δεν σημαίνει ότι πρώτα θα κηρύσουμε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και μετά θα προσπαθούμε να δούμε γιατί το κάναμε. Ευχαριστώ κυρία Παρβάνοβα. Η κυρία Γιανακουδάκη. Ένα λεπτό. Οι φήμες πάρα πολλές φορές είναι επικίνδυνες. Μερικές φορές οι φήμες ε, καταστρέφουν. <clears throat> Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις οι οποίες ε, δεν πήραν τις απαντήσεις που θα έπρεπε. Οι περισσότερες χώρες έχουν αναφερθεί στην ύπαρξη αυτού του ε, βακτηρίου. Έχουμε 22 νεκρούς σήμερα και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρξει σωστή και στενή συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές μια, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών σαν παράδειγμα θα πρέπει να ελέγχει και να πληροφορεί σωστά. Είμαστε αρκετά στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί είχαμε τρεις μόνο δηλωμένες περιπτώσεις. Αύριο όμως τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Θα πρέπει να βρούμε τις πηγές αυτής της μόλυνσης και να προστατεύσουμε το κοινό. Η Υπηρεσία Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών ε, κυκλοφορεί καθημερινές ενημερώσεις και μόνο αν είμαστε σωστά ενημερωμένοι μπορούμε να αποφύγουμε ε, περαιτέρω διάδοση της ασθένειας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Μινούτο. Ο κύριος Χουντής, ένα λεπτό. Μέσα σε έξι μήνες για δεύτερη φορά η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε αυτό που λέμε διατροφική κρίση με σοβαρά προβλήματα υγείας και ζωής ανθρώπων και συνανθρώπων μας. Εδώ κάτι δεν πάει καλά κύριε Επίτροπε. Τον Ιανουάριο είχαμε τις διοξίνες στη Γερμανία. Τώρα ξανά το βακτήριο πάλι στη Γερμανία. Η πρώτη περίπτωση καλύφθηκε ενώ ήταν γνωστή από μήνες. Η δεύτερη περίπτωση εύκολα μετατοπίστηκε στα αγκούρια της Ισπανίας. Πρόκειται περί προβλήματος αναγνωρισιμότητας, ιχνηλιασιμότητας και ανεπαρκούς ελέγχους σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης. στην πρώτη περίπτωση το γενάρη κύριε dalli μας είχατε πει μιλώντας για τις διοξίνες ότι θα πάρετε όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει πιο αυστηρή νομοθεσία στο σύστημα ελέγχου τροφίμων. προχτές δηλώσατε ότι δεν πρόκειται περί αυτού αλλά υπάρχει κάτι άλλο πρόβλημα δεν πρόκειται περί προβλήματος αναγνωρισιμότητας. η στάση της κομισιόν είναι σύγχυση κάλυψη πανικός στη συνέχεια με συνέπεια να έχουμε και να θρυνούμε σήμερα ζωές να θρυνούμε κρούσματα και να θρυνούμε συνέπειες στην αγροτική παραγωγή. Ευχαριστώ κύριε Χουντή. Για δύο λεπτά ο κύριος Γκαντίνη. Η κυρία Γκαντίνη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συζητούμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση και νομίζω ότι συνεχίσουμε να μπερδεύουμε σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικά πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να θέσουμε στο ίδιο επίπεδο τη ζωή κάποιων ασθενών και τα οικονομικά ζητήματα. Αυτό κάνουμε όμως. Επιπλέον, δεν μπορούμε μόνο με εντοπισμό αιτίων που δεν είναι αίτια να λύσουμε ένα πρόβλημα. Εάν έχω ένα φόνο και βάλω φυλακή έναν αθώο δεν σημαίνει ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Αυτό κάνουμε τώρα. Έχουμε μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση με μια υγειονομική κρίση, με μια διατροφική κρίση και εντοπίζουμε ένοχους που δεν είναι οι ένοχοι, δημιουργώντας, δημιουργώντας και άλλα θύματα δεν ε, κατέβηκαν στους δρόμους μόνο οι Ισπανοί Γεωργοί. Και στην Ιταλία σε λίγο βγαίνουν στους δρόμους στο Μιλάνο και στη Λατίνα οι Ιταλοί Γεωργοί που είναι ε, παραγωγή κυπευτικών, πετάγοντας στους δρόμους τα κυπευτικά τους, δίνοντας τον κόσμο κυπευτικά για να δείξουν ότι τα κυπευτικά είναι υγιής διατροφή. Ας μην επιβάλλουμε στους Γερμανούς κατανοητές διπλή βλάβη, να χάσουν τρόφιμα που είναι απαραίτητα για την υγεία και την διατροφή τους. Να σας δώσω κάποια στοιχεία που θα έπρεπε να μας κάνουν να σκεφτούμε, ιδίω στις αρχές όταν δίνουν πληροφορίες που δημιουργούν πανικό και ε, ανησυχίες. Στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Το 43% των Ιταλών όταν υπάρχει κρίση τροφίμων αποφεύγει να τρώει τρόφιμα που αναφέρονται για κάποιο χρόνο. 13% τα αποκόπτουν από τη διατροφή τους. Ξέρετε γιατί μιλάμε, ξέρετε πώς επηρεάζουμε την διατροφή ε, ατόμων. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να σκεφτεί μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσει η ρήτρα ε, κατεπήγοντος, ευρωπαϊκής κρίσης για την ε, κατάσταση στην ευρωπαϊκή διατροφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκαρντίνη. Η κυρία Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τάλη, εσεί και οι συνάδελφοί σα στη Γενική Διεύθυνση Υγεία, κάνατε τα πάντα σωστά. Αυτό δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμω για τι γερμανικές αρχές. Το ελάχιστο που πρέπει να πούμε είναι ότι υπήρξε ένα χάος επικοινωνίας. Για να μην τα πούμε τίποτα πιο σοβαρό. Το ότι το Υπουργείο Δημόσια Υγεία στην Γερμανία δεν θεώρησε ότι πρέπει να μεταβεί στο Λουξεμβούργο σε μια διάσκεψη των Υπουργών Υγεία που το κύριο θέμα ήταν ακριβώ αυτό, καταδεικνύει ότι δεν έχει ιδέα περί τίνο πρόκειται στην Ευρώπη. Αγνοεί τα προβλήματα ή εμπλήγεται μόνο σε ε, πολιτική κομματική μόνο. Ε, είπε, οι γερμανικές αρχές νόμιζαν ότι μπορούσαν να αρνηθούν τη συνεργασία των εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονό ότι οι εμπειρογνώμονε αυτοί μόλις τρει μέρε είναι στη Γερμανία είναι σκανδαλώδε επίση. θα πρέπει να το επικρίνουμε. Ταυτόχρονα μας που να πούμε αγαπητοί συνάδελφοι είναι υποχρέωση μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν να προειδοποιήσουμε τους καταναλωτέ όταν έχουμε ένα επικίνδυνο τρόφιμο στην αγορά. Και σα το λέω, εάν υπάρχουν βακτηρίδια σε ε, ένα αγγούρι σε σαλάτες ε, που δεν οδηγούν στο θάνατο είναι καλύτερο βέβαια αλλά είναι επίσης κακό και στα αγγούρια και στις σαλάτες υπήρχαν βακτηρίδια όχι τα ίδια αλλά υπήρχανε θα πρέπει, όταν υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, θα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί. Γιατί στην έγκαιρη προειδοποίηση θα πρέπει να κατονομάζεται, όπως ξέρετε, και το προϊόν και το όνομα του παραγωγού. Και θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει στο, στο μέλλον. Θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοπριά, θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι παραγωγής απαράδεκτες και θα δούμε ποιος έχει τι υποχρεώσεις σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ροτμπέραν. Το λόγο George Lyon. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πραγματική κρίση αυτή που έχουμε. 23 νεκροί. Πάνω από 2.000 ασθενείς. Ολόκληρες αγορές σε αναταραχή 300 εκατομμύρια ευρώ απώλειες καθημερινά για τους παραγωγούς και κρίση μεταξύ Γερμανίας και Ισπανίας, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Τρει εβδομάδε όμω μετά που ξεκίνησε η κρίση αυτή δεν ξέρουμε ποια είναι η πηγή μόνο τη. Η Υπουργέ Ντάλη θέλω να μου διαβεβαιώσετε σήμερα ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ανείχνευση της πηγής των βακτηριδίων αυτών. Γιατί αν δεν βρούμε τη πηγή δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε να ε, οικοδομούμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επίσης, όταν ξεπεράσουμε την κρίση, ποια είναι τα μέτρα που θέλετε να πάρετε για να σταθερόπιστε την ε, αγορά και να ξανακερδίσετε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επίσης, τρίτον, ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε για να δώσετε μια αποζημίωση σε εκείνους τους παραγωγούς που λόγω αυτής της κατάστασης έχουν καταστραφεί. Επίσης, θέλω να υπάρχει μια έρευνα το τι δεν πήγε καλά, γιατί μόνο αν το ξέρουμε μπορούμε να κλείσουμε τα κενά αυτά. Ευχαριστώ η Ελίζαπετ Κόστιγκαν για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, η υγειονομική πτυχή της κρίσης αυτής είναι τραγική πραγματικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Είναι απαραίτητο οι ε, παθόντες να βοηθηθούν και να ανοιχθούν όλα τα μέτρα για να αποφύγουμε περαιτέρω διεύρυνση της μόλυσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι υπάρχοντες πόροι. Τη κρίση της διαχείρισης ε, ανά την Ευρώπη ε, δείχνει ότι δεν είναι πολύ επαγγελματική η προσέγγιση. Υπήρχαν πρόορες αλληλοκατηγορίες, πράγμα που δεν βοήθησε παρά μόνο να οδηγεί στην πλήρη σύγχυση των παραγωγών των καταναλωτών. Για τους λόγο παραγωγούς υπάρχουν τεράστιες απώλειες εισοδήματος. Στη Γερμανία οι ε, αγορές ε, φρέσκων απορροκευτικών μειώθηκαν κατά 75% και αυτό σε πλήρη εποχή των προϊόντων αυτών. Ο, από όλα αυτά βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρη σήμαση των προϊόντων όσον αφορά την προέλευσή τους και τον έλεγχό τους. Ο καταναλωτής έχει το δίκιο να ξέρει από πού προέρχονται τα προϊόντα που καταναλώνει. Αυτό ισχύει και για την ε, πώληση σε ε, σούπερ μάρκετ αλλά και για την πώληση σε ε, εστιατόριο και άλλα γαστρονομικά κέντρα. Θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να ξαναξεκινήσουν οι πωλήσει των απορροκυπευτικών και να ενθαρρυνθεί επίσης πάλι το εμπόριο με τρίτες χώρες. Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν την καταστροφή χωρίς να φταίνει για τίποτα θα πρέπει η Κομισιόν να βοηθήσει μέσω παραδείγματο χάρη κινήτρων από το από το Ταμείο Γεωργίας. Έχει δίκιο ο Πέτερ Λίζε. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να ε, μετρηθεί σε χρήματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους που ε, βρέθηκαν στην κατάσταση αυτή χωρίς να φταίνει για τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κώστιγκερ. Η κυρία Γκασία Πέρες για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι θέλουμε η γερμανική κρίση διατροφής να κλείσει το σύντομο το δυνατό. Πρέπει να θυμηθούμε τα θύματα και ελπίζω ότι όταν διορθωθούν τα αρχικά λάθη θα βρούμε την αιτία της ασθένειας για να καθησυχάσουμε όλους. Ωστόσο, η υγειονομική παράμετρος της κρίσης δεν πρέπει να μας κάνει να γνωρίσουμε την οικονομική διάσταση του θέματος. Ο κλάδος ε, των οπωροκευτικών στην Ισπανία υπολογίζει τις ζημιές σε 200 εκατομμύρια ευρώ, ζημιές που προέρχονται από, τους μοιραίους, ε, από τα μοιραία κάθε επικοινωνία που γνωρίζουμε, παρότι ο κλάδο συνεργάστηκε απόλυτα με τι αρχέ τη χώρα μου. Κύριε Επίτροπε, η ανιχνευσιμότητα στην προέλευση λειτουργήσε. Αλλά πόσο χρόνο χάσαμε πηγαίνοντα στην προέλευση, κοιτάζοντα την γεωργική παραγωγή, ενώ αγνοούσαμε άλλε μορφέ μόλυνση στον προορισμό, όπω την επεξεργασία τη διανομή. Γιατί η Κομισιόν επικρότησε βεβαιασμένε πληροφορίε από τη Γερμανία, δεν υπήρξε συντονισμός επίτροπε. Οι μονομερείς ε, αποκλεισμοί των συνόρων για ισπανικά προϊόντα είναι απόδειξη των ε, ελλείψεων της, της αντιμετώπισης της κρίσης στην Ένωση. Ζητώ από την Επιτροπή να ενεργοποιήσει αμέσως όλους τους μηχανισμούς για να αποζημιωθεί ο ευρωπαϊκός και ισπανικός κλάδος και οικονομικά και από την οπτική γωνία της εικόνας του στον καταναλωτή. Μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρχουν και άλλα σχετικά μέτρα. αβάσιμες καταγγελίες, αυτοσχεδιασμοί, έλλειψη συντονισμού, απόλυση εκατομμυρίων, επίθεση στην τιμή και την αξιοπιστία του κλάδου. Δεν είναι αρκετά για να ζητήσουμε ευθύνε. Ευχαριστώ κύριε Γκαρσία Πέρε. Νομίζω ο συνάδελφος Πούλσεν λείπει. Κυρία Μαγκίνες, λοιπόν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Ντάλη, ευχαριστούμε για τα μετρημένα σχόλιά σας στο ξεκίνημα της συζήτησης. Τα λιγότερα, ωστόσο, μετρημένα λόγια για το κόστος στην ανθρώπινη ζωή και στους, ε, και στους παραγωγούς. Πρόκειται για, μια, για την πιο σοβαρή, μια εξαιρετικά σοβαρή κρίση. Ξέρουμε ότι πλήττει ένα κομμάτι της Ένωσης, αλλά δεν είναι γερμανικό, είναι ενωσιακό πρόβλημα. Το σύστημα υπάρχει για να αναζητείται η αιτία και να αντιμετωπίζονται οι συνέπειές της. Φοβούμαι ωστόσο ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα, και δεν λειτουργήσαν σωστά όλα τα τμήματα του συστήματος η έγκαιρη προειδοποίηση, από ό,τι κατάλαβα, ξεκίνησε στις 22 Μαΐου. Οι, ε, οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες, ωστόσο, και αυτό με ενσυχεί, έφτασαν στη Γερμανία προχτές, 5 Ιουνίου. Γιατί τέτοια χρονική απόσταση. Αυτό πρέπει να το δούμε. Έχουμε, όπως βλέπω, βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού 178 ε, του 2002, τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων Όλοι λένε ότι είναι κρίση. Και εσείς είπατε ότι είναι κρίση. Κρίση που εξελίσσεται, αυξάνεται. Προτείνω λοιπόν τώρα η Ένωση να επικαλεστεί το περιεχόμενο του κανονισμού αυτού και να δημιουργήσει αυτή την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων. Το πιο ανησυχητικό είναι η μνήα, η, αναφορά, η αναφορά ευθύνη για συγκεκριμένα ε, κυπευτικά και μετά τους λέμε όχι για να θω αυτά. Αυτό είναι σοβαρότατο πρόβλημα και στην ασφάλεια των θύμων και στον έλεγχο. Κύριε Ντάλη, ξέρω ότι θέλετε να υπάρξει συμφωνία, πιστεύω ωστόσο ότι είναι καιρός τώρα να ξεκινήσετε αυτή τη μονάδα κρίσης. Θα ήθελα σχόλιά σας στο τέλος. Η κυρία Ρόντουστ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επιτροπή. Εγώ προέρχομαι ακριβώ από την περιοχή της ε, Γερμανία, όπου υπάρχει αυτό το μακτεριδιό. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να σταματήσει η εξάπλωσή του. Από τα μέσα Μαΐου μέχρι χθε είχαμε 1733 ασθενεί και 33 πέθαναν. Απεβίωσαν. Οι κατάσταση κλινικέ είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Δεν υπάρχουν πια ε, κλίνε στι μονάδε και ζητούν πλάσμα αίματος. Για μένα αυτό σχετίζεται με την ε, ανάληψη ευθυνών. Έγινε ανάλυση διαφόρων τροφίμων χωρίς να βρεθεί μέχρι στιγμής τίποτα. Από όσο καταλαβαίνω εγώ, τρόφιμα υψηλής ποιότητα θα πρέπει να είναι υγιή και να φτάνουν ελεγμένα στο εμπόριο. Εδώ έγιναν κάπου τεράστια σφάλματα και για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά κενά. Στην κατάσταση αυτή να πούμε ότι γνωρίζουμε το... την προέλευση χωρίς να υπάρχουν εργαστηριακά αποτελέσματα δεν επιτρέπεται. Κατανοητός ο πανικός. Παρ' όλα αυτά όμω δεν θα πρέπει να φτάσουμε στο κυνήγι των μαγισσών γιατί αυτό σημαίνει ότι οδηγούμε σε καταστροφή πολλούς παραγωγούς σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνουμε ε, αλληλέγγυοι και να βοηθούμε οι μεν τους δε όταν υπάρχει ανάγκη. Σε ιατρικό επίπεδο θα πρέπει δηλαδή όλοι οι εμπειρογνώμες να κάτσουν από το ίδιο τραπέζι και οικονομικά να βοηθηθούν εκείνοι που αθώοι κατα... Δύο λεπτά η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτον, να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια προς, τα, προς την οικογένεια των θυμάτων. Κύριε Επίτροπε, η ανακοίνωση των υγειονομικών ζητημάτων στην κοινή γνώμη είναι δύσκολο, λεπτό ζήτημα και πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Όχι, ο στόχος δεν πρέπει να είναι να βρεθούν ένοχοι. Εδώ έγιναν τεράστια λάθη με τις παράτολμες και βεβαιασμένες κατηγορίες περιφερειακών υπευθύνων κατά ε, συγκεκριμένων ατόμων που δημιούργησαν κοινωνική αναταραχή και σοβαρότατη ανεπανόρθωτη οικονομική κρίση. Ούτε και η Κομισιόν αντιμετώπισε το ζήτημα σωστά. Ρωτώ, πότε έγινε, πότε εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα, έγινε, χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 3 του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που υποχρεώνει τους κινδύνους να ε, κοινοποιούν αμελητή τους κινδύνους σε 48 ώρες. Τηρήθηκε το άρθρο 8 του ίδιου κανονισμού που υποχρεώνει την Επιτροπή να επαληθεύσει κατά πόσον οι πληροφορίες ε, που παρέχονται είναι πλήρεις και έχουν πολύ σωστή νομική βάση. Προφανώς εμφανίστηκαν οι σοβαρές ελλείψεις στον κανονισμό αυτό και οι σοβαρέ ελλείψει στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που πρέπει να αναθεωρηθεί. Επιπλέον, να ορίσουμε σαφώ τι διαδικασίε αντιμετώπιση κρίση από πλευρά των αρμοδίων αρχών. Να αναθέσουμε συγκεκριμένους ρόλους στους υπεύθυνους της αλυσίδας διατροφής. Αυτό είναι και ο λόγος της λιχνευσινότητας. Να αποφύγουμε η προστασία υγείας να χρησιμοποιείται για, ε, για εμπορικά εμπόδια. Να, να αποζημιώνουμε αυτούς που άδικα πλήττονται. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι ούτε τα αγκούρια, ούτε η σόγια η αιτία, αλλά ο, παθογεν, ο παθογόνος παράγοντας όπως αναφέρθηκε. Είναι Το όμικρον 181 H4 του E. coli που δημιουργεί ε, το κρούσμα. Ωστόσο κύριε Επίτροπε πρέπει να αφήσουμε τους επιστήμονες να δουλέψουν, να βρουν το προϊόν, να, να ζητήσουν την αλυσίδα διαφοροφή και την χρησιμοποίηση και επεξεργασία των τροφίμων και στη διανομή και στην ε, ε, χρησιμοποίηση. Ο κύριος Περέγιο Ροντρίγκες, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτά που κάνουμε εδώ ή στην Ένωση δεν θα φέρει πίσω στη ζωή τους νεκρούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ούτε θα μειώσουμε τη, τα προβλήματα των ασθενών. Δεν ξέρουμε την αιτία. Ξέρουμε όμως κάτι και πρέπει να το πούμε. Υπήρξε αμέλεια, πολιτική αμέλεια και αμέλεια της γερμανικής κυβέρνησης. Δεν μπορεί να λέμε ότι το, να, να, να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση λέγοντας ότι το Αμβούργο είναι κάπου αλλού. Η κυρία Μέρκελ με υπεροψία αντιμετώπισε την κατάσταση, δεν προχώρησε σε, σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης. Αν είχε προχωρήσει πιο προσεκτικά δεν θα είχαμε ε, τα προβλήματα. Ε, ε, ε, έπληξε ένα κράτος και, μια, και έναν οικονομικό κλάδο δημιούργησε σοβαρότατα προβλήματα στην οικονομία και συγκεκριμένη περιοχή και ζητώ να πάμε στο Συμβούλιο και να αποφασιστεί το Συμβούλιο πλήρης αποζημίωση των θηγέντων. Ζητούμε να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχου και να απαιτηθεί ευθύνη τη κυρία Μέρκελ να απατηθεί να λειτουργούν με μεγαλύτερη, ε, με μεγαλύτερη προσοχή. Δεν μπορεί να πούμε ότι άλλο κρατήριο του Αμβούργου δεν έχουμε εμεί ευθύνη. Δεν μπορεί ε, να χρησιμοποιείται το ομοσπονδιακό σύστημα για να απεμπλέκονται οι ευθύνε ορισμένων. Ή θα θα έπρεπε η κρίση αυτή να μην μας ξεφύγει από τα χέρια και αν είχε δράσει σωστά η Γερμανία θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετική ε, κατάσταση, διαφορετική εξέλιξη. Κύριε Επίτροπε, το ζητούμε από εσά και από το γερμανικό κράτος μεγαλύτερη ευθύνη και καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. Η, κυρία Τελάνγκε, δύο λεπτά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντάλη που είναι ανάμεσά μας σήμερα θα προτιμήσα να είναι αλλού βέβαια, να πηγαίνει στη Ρωσία με το αεροπλάνο για να τους πείσει ότι είναι άδικη η απαγόρευση εισαγωγής ε, ευρωπαϊκών οποροκυπευτικών. Θέλω να ευχαριστήσω παρόλα αυτά ε, τον Επίτροπο για την ενημέρωση την οποία μας έκανε. Ενημέρωση βέβαια η οποία ήταν ε, μέχρι τώρα θα έλεγα αποτυχημένη. Υπήρξε μια συνέντευξη που δόθηκε από τον αρμόδιο επίτροπο αλλά ήδη όταν δόθηκε η συνέντευξη είχαν κυκλοφορήσει τρεις ιστορίες είχαν καταδικαστεί ακόμα και τα Ολλανδικά αγκούρια, κάναμε τεράστιες ποσότητες τεστ και δεν βρέθηκε φυσικά τίποτα. το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε αλλά υπήρξαν προβλήματα επικοινωνίας. Στη Γερμανία υπάρχει μια ολόκληρη σειρά αρμοδίων αρχών, Ινστιτούτων, ερευνητικών κέντρων και μεταξύ τους υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση και έγιναν πολλές λανθασμένες ανακοινώσεις από πλευράς των γερμανικών υπουργείων, τα οποία μάλιστα παρενέβησαν και σε τομείς οι οποίοι δεν ήταν αρμοδιότητά τους. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους Γερμανούς για να έχουμε κάποιες περισσότερες εξηγήσει για το γιατί πήγαν τα πράγματα τόσο άσχημα. Θα συναντηθείτε και με τους Υπουργούς Γεωργίας κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ποσό ε, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιείται σε περίοδους κρίσης όπως το είχαμε κάνει στο παρελθόν για τον γαλακτοκομικό τομέα. την εβδομάδα χάνονται 80 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τους Ολλανδούς παραγωγούς. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες πήγαιναν πολύ καλά και οι οποίες τώρα απειλούνται με καταστροφή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και οι Υπουργοί Γεωργίας. Ευχαριστώ ε, κυρία Ντελάνγκε. Η κυρία Ζαμπόρσκα έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, καλωσορίζω την συζήτηση αυτή. Το πρόβλημα το βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες. Πρώτον, από την προέλευση της ασθένειας. Ποια είναι η αιτία της, δημιουργώντας και την σωστή θεραπεία. Μία εταιρεία, μία φαρμακευτική εταιρεία πρότεινε, όπως διαβάζω, κάποια θεραπεία. Πιστεύω ότι έγιναν πολλά λάθη στην πληροφόρηση. Πληροφόρηση των πολιτών κυρίως. Αν πείτε στους πολίτες μην αγοράζετε ένα τρόφιμο σήμερα γιατί μπορεί να μην είναι υγιές, αυτό είναι μια τελείως ανεύθυνη πράξη. Η ενημέρωση των πολιτών πρέπει να είναι υπεύθυνη με ενιαία εκστρατεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να λέμε στους πολίτες τι να κάνουν το πρωί και τι να κάνουν το βράδυ. Αν τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής προφανώς, προσωπικούς, αν πλένουν τα τρόφιμα, τα μαρούλια, αν τα μαγειρεύουν σωστά. Αυτοί είναι βασικοί κανόνες που ούτως ή άλλως θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ή να προλάβουν τέτοιες επιδημίες. Αυτή θα πρέπει να είναι λοιπόν η αλλω θα μπορουσαν να αντιμετωπισουν η να προλαβουν τετοιε επιδημιε αυτη θα πρεπει να ειναι λοιπον η καμπανια που θα πρέπει να, στην οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να λέμε στους πολίτες βασικούς κανόνες υγιεινής. Δηλαδή η προσωπική συμπεριφορά μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες κρίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζαμπόσκα. Διαδικασία Κατσουιάη. 21 αιτήματα παρεμβάσεως ε, λάβαμε μετά από αυτή τη μακρά εξαιρετικά δικαιολογημένη συζήτηση. Πλην όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα να δεχθούμε όλα τα αιτήματα παρέμβαση. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που δεν θα καλέσω στο βήμα. Πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο αλλιώς ε, καθυστερούμε τις υπόλοιπες συζητήσεις. Πρώτη παρέμβαση. Σικίερσκι. Είναι σημαντικό Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και για τον πληθυσμό τον γενικό και για τους ε, διαφορετικού τύπου κίνδυνοι και για τους παραγωγούς των προϊόντων τα οποία αμφισβητούνται σήμερα. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής και της ποιότητας ε, και της υγιεινής του, το οποίο πρέπει να είναι ικανοποιητικό, φέρεται να είναι ικανοποιητικό. Συνεπώς ε, ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων δεν πρέπει να χρειάζεται τόσος χρόνος για να βρούμε ποιες είναι οι πραγματικές πηγές της μόλυνσης δεν θα πρέπει να ανακοινώνονται πληροφορίες όταν δεν είναι επιβεβαιωμένες που οδηγούν σε τεράστιες οικονομικές απώλειες. Τα συλληπιτήριά μου φυσικά στα θύματα και στις οικογένειές τους προφανώς, αλλά να μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα οικονομικά θύματα. Εδώ το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε έχει άμεση σχέση με το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι κάτι το οποίο δεν έχει μόνο σχέση με, το, με τα τρόφιμα, αλλά έχει σχέση και με την οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε με μία μορφή επιδημίας, όπως ξεκαθάρισε ο κύριος Επίτροπος Ντάλι. Στην ουσία, αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε τις πραγματικές αιτίες, προσπαθήσαμε να βρούμε ποιος φταίει. Τρεις εβδομάδες μετά δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Η αρχή της πρόληψης εφαρμόζεται βέβαια, αλλά παρόλα αυτά, χωρίς να χρησιμοποιηθούν επιστημονικές αποδείξεις και τεκμηριώσεις, καταδικάστηκε η Ισπανία η οποία δεν είχε καμία σχέση φυσικά και η παραγωγή των προϊόντων της με το ξέσπασμα της μόλυνσης. Αυτό οδήγησε σε μια καταστροφή στον τομέα της παραγωγής των οποροκυπευτικών στη χώρα μου. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε ε, περισσότερες απαντήσεις κύριε Επίτροπε. Ε, η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αλλά δεν φταίει η Ισπανία γι' αυτό και γι' αυτό πρέπει να μας αποζημιώσετε για τη ζημιά που μας προκαλέσατε. Κύριε Ντουρό, κύριε Επίτροπε, διευκρινίσατε ότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό και θα πρέπει να το ε, ξεκαθαρίσετε αυτό ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα και μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού. Νομίζω ότι το μήνυμα που δόθηκε ήταν ιδιαίτερα, ε, προκάλεσε μια πολύ μεγάλη σύγχυση και στο σύνολο του κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά στην Ισπανία και στη Γερμανία. Ανάμεσα στη διαφάνεια και στις πρόορες ενημερώσεις είναι μια δύσκολη ισορροπία. Αλλά νομίζω ότι η αρχή της πρόληψης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πρέπει να διαδίδουμε ατεκμηρίωτα στοιχεία χωρίς κανένα λόγο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε και τι αποζημίωση θα δοθεί σε αυτούς οι οποίοι εφήγησαν. Αυτά θα συζητήσετε σήμερα το απόγευμα. Αλλά φυσικά αυτοί που μας απασχολούν περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι υπέκυψαν, είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν. Το θέμα πάντως της ανιχνευσιμότητας είναι ένα θέμα στο οποίο πολλά μένει να γίνουν. Έχουμε 22 νεκρούς αυτή τη στιγμή και άνω των 2.000 ασθενών ε, μετά το ξέσπασμα της επιδημίας σε σκερίχια κόλλη. Θα πρέπει φυσικά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας σε αυτούς που έχασαν τους συγγενείς τους και να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στους υπολείπους. Θα πρέπει να έχουμε τρόφιμα τα οποία να είναι ποιοτικά και να είναι φυσικά ανιχνεύσιμα. Οι απαντήσεις ε, φαίνεται ότι δεν ήταν ικανοποιητικές μέχρι τώρα και γι' αυτό υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Υποφέρουν οικονομικά οι γεωργοί, ενώ τα προϊόντα τα οποία παράγουν είναι απόλυτα ασφαλή. Βέβαια να υπάρξει επίσης και περισσότερη ψυχραιμία. Οι εθνικές κυβερνήσεις πάρα πολύ γρήγορα απέδωσαν ευθύνε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τέτοιου είδους ε, φήμες ε, είχαν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν. Πριν υπάρξουν απαγορεύσεις περαιτέρω θα πρέπει να ελέγξουμε τα γεγονότα. Η κυρία Τερέσα Χιμένες. Αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι τα θύματα. Δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε τα θύματα τα οποία έχουν υπάρξει. Θα πρέπει μέσα από τη διαδικασία αυτή να βγούμε ενδυναμωμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε τους υπευθύνου και δεν μπορώ παρά να καταγγείλω και εγώ τις γερμανικές αρχές οι οποίες καταδίκασαν τη δική μου χώρα και ιδιαίτερα του συνεταιρισμού της Αλμέρια που είναι θα έλεγα πρότυπο εκμετάλλευσης γεωργικών προϊόντων και παρόλα αυτά οδηγήθηκαν σε τεράστιες απώλειες θέσεων απασχόλησης που διαρωτώνται γιατί συνέβη αυτό το οποίο συνέβη και ποιο θα είναι το μέλλον τους. Συνεπώς, ελπίζω οι εμπειρογνώμονες να μας δώσουν μια απάντηση το ταχύτερο δυνατόν. Παρακαλώ όταν συναντηθείτε με το Συμβουλίο να του ζητήσετε να ληφθούν οικονομικά μέτρα απόσβεσης των ζημιών ε, και για τους καταναλωτές αλλά κυρίως για τους παραγωγούς. Είμαστε αγανακτισμένοι αλλά ελπίζουμε κιόλας. Απαιτείται περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία, λέει ο κ. Ιδάλγο. Κατασυκοφαντήθηκαν οι παραγωγοί στην Ισπανία. Οι Γερμανοί μέχρι τώρα δεν έχουν προχωρήσει σε καμία μορφή, σε καμία μορφή αποζημίωσης των παραγωγών στην Ισπανία. Ο τρόπος με τον οποίο η Μέρκελ αντιμετωπίζει τις νότιες χώρες είναι απαράδεκτος δεν έχει αξιοπιστία. Ευχαριστώ κύριε Μάσιπ. Ο κύριος... Ευχαριστώ κύριε Μάσιπ. Ο κύριος Στάς έχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι κύριε Επίτροπε. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που έγιναν. Έλλειψη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε γερμανικό επίπεδο, το είπαν και οι γερμανοί συνάδελφοι, έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, χρειάζεται πολύ σοβαρό εθνικό σύστημα ελέγχου και αυτό πρέπει να συμβεί όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλα τα κράτη-μέλη. Δείχνουμε τώρα τη Γερμανία, αλλά δείτε τι γίνεται στις χώρες μας. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να το δούμε παντού. Εσωτερική έλεγχη στα κράτη-μέλη είναι επαρκώς ισχυρή για να αντιμετωπίσουν τέτοιες ε, καταστάσεις. Υπάρχουν συστήματα ελέγχου που λειτουργούν, υπάρχει έλλειψη συντονισμού και αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα των κύριων, του κύριου Λένε της κυρίας Ροτ Μπέρεντ. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε στη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας για την αποζημίωση όσων επλήγησαν οικονομικά. Πρόεδρε. Στην κρίση φαίνεται η αποτελεσματικότητα. Εδώ δεν φάνηκε. Είπε ο Επίτροπος ότι οι υποψίες για τα ισπανικά αγκούγια δεν επιβεβαιώθηκαν. Όχι κύριε Επίτροπε. Επιβεβαιώθηκε ότι οι υποψίες ήταν αβάσιμες. Επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν 23 νεκροί και ότι υπήρξε τεράστια βλάβη του κλάδου στην Ισπανία. Επιβεβαιώθηκε ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει αυτό που δεν έκανε μέχρι τώρα. Με αποφασιστικότητα σε κάθε επίπεδο αντιμετώπιση της κρίσης και αποφυγή αθεμελίωτων κατηγοριών που, δίνουν, που οδηγούν σε τεράστιες οικονομικές συνέπειε για κάποια κράτη, την Ισπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποζημιώσει αμελητή τους θυγέντες και να αποκαταστήσει στα ισπανικά προϊόντα την ε, βεβαιότητα ότι είναι ασφαλή και καλής ποιότητα προϊόντα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζούντιτ Μέρι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, βρισκόμαστε εν μέσω της κρίσεως. Νομίζω ότι έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε από το να ψάχνουμε ενόχους. Πιστεύω ότι πρέπει να λύσουμε καταρχάς την κρίση και κατόπιν να δούμε την πρώτη προτεραιότητα που έχουμε. Μία θεραπεία για τους ασθενείς. Να βρούμε την πηγή της μόλυνσης και να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Αυτά είναι, αυτή είναι η στόχη. Να ενημερώνουμε τους καταναλωτές και τους ασθενείς. Να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα όλων. Κατόπιν να δούμε πώς θα χειριστούμε κρίσεις εν γέννη. Παρεμβαίνουν υπερβολικά κάποιες αρχές, παρεμβαίνουν λιγότερο από ό,τι πρέπει κάποιες άλλες. Και πρέπει να συζητήσουμε στο Συμβούλιο πώς θα αντιμετωπίζονται στο μέλλον οι κρίσεις και από ποιους. Νομίζω ότι η κρίση δείχνει πως υπάρχουν μεταξύ των χωρών πολύ μεγάλες διαφορές κατόπιν. Χρειάζεται αποζημίωση όσων άδικα εθίησαν. Η κυρία Αγγέλικα Βέρτμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οπωσδήποτε τα συστήματα μας πάνε προς τα θύματα. Για να προστατευτεί όμως το σύνολο του πληθυσμού οι αρχές έχουν την υποχρέωση να τους προστατεύσουν. Τη είπα, υπάρχει ένα έγκαιρο σύστημα προειδοποίηση. Αυτή τη στιγμή όμω εμείς έχουμε πάνω από 2.000 ε, ασθενεί και 20 νεκρός. Θα πρέπει να ε, δούμε ε, κατά πόσο πραγματικά αυτό προέρχεται από τα αγκούρια. Δεν έχει καμία σχέση όμως το αγκούρι με αυτά τα βακτηρίδια που προέρχονται από τα απορρίμματα. Και βρίσκω πολύ άσχημα που το Συμβούλιο απουσιάζει από όλη τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Bogosław Σόνικ. ευχαριστώ, λέει ο κύριο Σόνικ, που μου δώσατε το λόγο σε μια συζήτηση την οποία βρίσκω ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν μεγαλύτερη ανταπόκριση από του μηχανισμού τη. Μόνο μια τέτοια ανταπόκριση θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιου είδους επιδημίες από το να εξαπλωθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να έχουμε επίσης μεθόδους οι οποίες να είναι πλήρως ανεξάρτητες από τις δημόσιες διοικήσεις και θα πρέπει να είναι μέθοδοι που διασφαλίζουν τη μη εξάπλωση του πανικού στους καταναλωτές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς ο πανικός προκλήθηκε. Οι συνέπειες είναι πλέον γνωστές και υπήρξαν τεράστιες απώλειες ε, ε, οικονομικές για τους παραγωγούς. Θυμίζω ότι οι τιμές στα οποροκυπευτικά στην Πολωνία έπεσαν κατά 60% τις τελευταίες εβδομάδες. και ταυτόχρονα σε αντίστοιχες ε, ζωνόσους στον τομέα της παραγωγής χείριου κρέατος δημιουργήθηκαν αντίστοιχα προβλήματα στο παρελθόν. Κύριε Πρόεδρε, σε τέτοιε περιπτώσει η ελεγγύη πρέπει να λειτουργήσει. Δεν ε, πρέπει να αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν ε, είναι συνήθες, δεν είναι κανονικό να πηγαίνουν οι Γερμανοί και να αφήνουν στην Ευρώπη την ευθύνη. Ήδη από την πρώτη συνέντευξη τύπου φάνηκε ότι ε, ε, ε, αυτό ήταν λάθος. Δεν είναι σωστό να κατηγορούμε χωρίς αποδείξεις, χωρίς επικοινωνία. Δεν είναι συνήθες οι αρχές επικοινωνίας στις κρίσεις να αγνώνται με τέτοιο τρόπο. Γι' αυτό περάσαμε από την κρίση στην ψύχωση. Οι φήμες, το κυνήγι μαγισσών έβλαψαν σημαντικότατα όσο και η ίδια η ασθένεια. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, πρέπει να επαναποκατασταθεί. Για να μην επανέλθει το δράμα αυτό χρειαζόμαστε να μάθουμε πρώτον να βελτιώνουμε καλύτερα την ε, διασυνορική ανεχνησιμότητα και να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή μονάδα επικοινωνιών και διαχείριση κρίσεων για να μάθουμε τα μαθήματα από αυτή τη αποτυχία και να μην έχουν πεθάνει άδικα 21 άτομα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Δέκα συνάδελφοι μίλησαν ήδη μέχρι εδώ. Ζητώ συγγνώμη από τους άλλους 12 που δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν. Κύριε Επίτροπε, έχετε τώρα το λόγο για να συνοψίσετε. Δύσκολο βέβαια να συνοψίσετε μια τόσο πλούσια συζήτηση, αλλά σας ε, προκαλώ. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που πήραν μέρος στην συζήτηση. Δεν έχω τον χρόνο φυσικά να αντιδράσω σε όλες τις επιμέρους ερωτήσεις και σε όλα τα ενδιαφέροντα σχόλια τα οποία κατατέθηκαν, αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι λάβαμε, σημειώσαμε τις απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν από πλευρά σας. Όπως σας είπα σήμερα το απόγευμα θα είμαι στο Συμβούλιο Γεωργίας και αύριο το πρωί θα είμαι στο Βερολίνο και θα πάρω μέρος σε μια συντονιστική συνάντηση ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας και τους δικούς μας εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την διάδοση ε, του προβλήματος. Αυτός είναι ο βασικός στόχος συγκεντρώνουμε την ε, πρόσοχή μας στην επιτάχυνση των διαδικασιών ε, εντοπισμού των αιτιών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμείς από το τέλος Μαΐου έχουμε κινητοποιηθεί πλήρως. Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν κινητοποιήσει τα συστήματα ελέγχου, το ECDC, το οποίο έχει κινητοποιήσει με τη σειρά του επίσης και τις διαδικασίες ελέγχου των κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αμέσως από το ECDC να προχωρήσει σε επιστημονικές μελέτες και αξιολογήσεις με πάρα πολλές συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια προ ιατρούς, προς ασθενείς ε, και επίσης ε, δώσαμε και πολλές συστάσεις και συμβουλές οι οποίες κυκλοφόρησαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα στη σωστή τους προοπτική. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για όλους το να καθίσουμε και να καταδικάζουμε δεξιά και αριστερά. Αντίθετα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο κέντρο του προβλήματος και να διαχειριστούμε την κρίση. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην εκεί που κάνουμε, γιατί από τη μία θα πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται μόνο με συγκεκριμένες αποδείξεις, από την άλλη δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, μερικές φορές να λαμβάνουν παρακινδυνευμένες αποφάσεις σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες γιατί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πολλές φορές φοβούνται ότι εκ των υστέρων θα κατηγορηθούν για τις αποφάσεις αυτές. Μην το ξεχνάτε αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα τμήμα της διαχείρισης της κατάστασης που δεν πρέπει να αγνοούμε. Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο των πληροφοριών που κυκλοφορούν. Έχουμε ένα σύστημα στην Ευρώπη το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή στοιχείων με μεγάλη ταχύτητα και γι' αυτό ακριβώς εφαρμόζουμε και την αρχή της επικουρικότητας. Φτάνουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται στην πυραμίδα για να δούμε ποιες είναι οι πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να πάρουμε από την αρχή που προκαλείται το πρόβλημα και προσπαθούμε ε, σιγά σιγά ανεβαίνοντας προς τα πάνω με τους ελέγχους ε, στρώμα προς στρώμα θα έλεγα επίπεδο προς επίπεδο να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε σίγουρα συμπεράσματα. Η ταχύτητα είναι απαραίτητη και ε, φυσικά ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας της ζωής. Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε όσο παίρνουμε πληροφορίες με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της ενημέρωσης τουλάχιστον έχουμε συμφωνήσει ότι η ταχυτάτη ενημέρωση είναι βασικός στόχος της σωστής διαχειριστικής προσπάθειας. Είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν με αντίστοιχες κρίσεις ένα καλό σύστημα ενημέρωσης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μας έχει ένα δίκτυο θα έλεγα κέντρων όπου θα προέρχεται, από τα οποία θα προέρχεται η σωστή ενημέρωση Ήμουνα σε επαφή και με τους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έτσι ώστε η ενημέρωση να δίδεται εκεί όπου χρειάζεται. Θα προχωρήσουμε στη μελέτη λοιπόν την προσεκτικότερη όλων όσων έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Θα προχωρήσουμε σε έρευνες, σε αναλύσεις και μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι η διάδοση θα έχει πλέον σταματήσει τότε θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και στον τομέα της ενημέρωσης και στον τομέα των πρωτοκόλων και στον τομέα της σωστής ενημέρωσης γενικότερα. και σε ένα υστερότερο στάδιο θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι χρειάζεται για να βελτιώσουμε την επικοινωνία ανάμεσα στους Ευρωπαίους, στις ευρωπαϊκές χώρες. Εν πάση περιπτώσει πάρα πολλά θέματα τίθενται προς συζήτηση και στο δικό σας επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Το θέμα των αποζημιώσεων θα συζητηθεί σήμερα στο Συμβούλιο Γεωργίας και είμαι σίγουρος ότι ο συνάδελφός μου ο κ. Τσίολος κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να φροντίσει να βρεθούν τρόποι αποζημίωσης των γεωργών οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξ αυτού του θέματος που συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ολοκληρώνεται το θέμα αυτό και θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα